στις 19 έχει εξαντληθεί η ημερήσια διάταξη και θα είναι η ημερήσια διάταξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.